το Λάος και το Βιετνάμ. Ακολουθεί η συζήτηση σχετικά με πέντε ψηφίσματα για την Κίνα, μειονοτικά δικαιώματα και θανατική ποινή. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Ντεκέζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου έχει αποσύρει την υπογραφή της από το ψήφισμα για την Κίνα. Γιατί? Όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι δευτερεύον το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι είναι λιγότερο σημαντικό από τα εμπορικά συμφέροντα. Εμείς είμαστε στεναροί στην ε, δέσμευσή μας. Αλλά για να έχουμε κάποια πρόοδο στην Κίνα πρέπει να έχουμε ένα διάλογο. Το ψήφισμα αυτό το οποίο είναι αποσπασματικό και εμβαλωματικό δεν μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το διάλογο. Ασχολείται με τις θρησκευτικέ ε, εκστρατείες, με το Δαλάι Λάμα, με το Θιβέτ με όλα τα προηγούμενα και τωρινά κομμουνιστικά καθεστώτα. Δεν είναι ο τρόπος να ανοίξουμε μια πόρτα για την Κίνα. Το δράμα είναι ότι κλείνουμε ακόμα και τις μικρές πόρτες που παραμένουν ανοιχτές και δεν βοηθάει ούτε καν να σώσουμε τους Ουιγούρους και τους Θιβετιανούς που απειλούνται με εκτέλεση. Είναι απαραίτητο να έχουμε επαφές όχι μονάχα εμπορικές και όχι πολιτιστικές και μόνο, αλλά και μέσω των κοινών αξιών. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη προσεχού Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, στο θέμα της στρατικής ποινή και ζητώ από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να εξακολουθήσουν να θέτουν μέσα στα πλαίσια της νέας εταιρική σχέσης για την ε, Κίνα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Κίνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χίγκης για δύο λεπτά. Ε, ε, President. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υποστηρίζω τις εκκλήσεις για το, την κατάργηση θανατικής ποινής στην Κίνα και ιδίω όταν η θανατική ποινή χρησιμοποιείται για να τρομοκρατούνται οι μειονότητε, οι εθνοτικέ ομάδε και τα έθνη τα οποία διαβίουν μέσα στο κινέζικο κράτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Πολιτείε και άλλε δυνάμει σε παγκόσμιο επίπεδο παρόλα αυτά, όταν επικρίνουν τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, είναι ιδιαίτερα ήπιοι και όταν πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι σχεδόν ανύπαρκτη η επίκρισή τους. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές σχέσεις με τις κινέζικες εταιρείες και τη γραφειοκρατία η οποία ελέγχει το κινέζικο κράτος ώστε να υποφεληθούν από την αποτρόπαια εκμετάλλευση των εργαζομένων στην Κίνα. Η Κίνα είναι ένα γιγάντιος, ένας γιγάντιος τόπος σκλαβιάς εργασία σκλάβων, όπου εκατομμύρια εργαζομένων, δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένων ζουν μια φρικτή ζωή και οι ίδιοι και τα παιδιά τους πλήττονται από τις φρικτές συνθήκες στις οποίες ζουν. Οι εταιρείε πολυεθνικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ συμμετέχουν σε αυτόν τον τρόπο εκμετάλλευσης με στόχο να αυξήσουν τα υπερκέρδη τους. Το κινέζικο καθεστώς αυξάνει, δεν μειώνει την καταστολή και αυτή η καταστολή έχει οξυνθεί από τότε που το σταλινικό καθεστώς της Κίνας αποφάσισε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της οικονομίας της αγοράς για να αναπτύξει την κινέζικη οικονομία. Έχει αυξηθεί η καταστολή των δημοσιογράφων και των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρόσφατα ένα σοσιαλιστής συναδελφός μου εξεδιώχθη από την Κίνα. Ο Βίνσεντ Κόλερ ο οποίος είναι ο εκδότης ενός εντύπου για τους εργάτες στην Κίνα, εμποδίστηκε, του εμποδίστηκε να μπει στην Κίνα, τον απελάσαν από την Κίνα, γιατί ήταν αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξουν τα εργασιακά δικαιώματα στην Κίνα, θέλουμε να απολυθούν όλοι οι πολιτικοί ε, κρατούμενοι και ακτιβιστές ελευθερία του συνέρχεσαι και έκφραση, Διεθνή αλληλεγγύη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ολιγαρχικό γραφειοκρατικό καθεστώς που μοιάζει πάρα πολύ με το αντίστοιχο σύστημα στη Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Αντρική. Είναι ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι δεσμοί μας ενισχύονται με την Κίνα στον τομέα του περιβάλλοντος, του εμπορίου και οργάνωσε και τους περίφημους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι. Δυστυχώς πάει πίσω στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της. Καταστέλει με δύο τρόπο τις ειρηνικές διαδηλώσεις στο Θιβέτ πέρυσι και στο Σινκιάνγκ φέτος με εντελώς δυσανάλογη χρησιβίας. Όλοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διαδηλώνουν εναντίον των κυβερνήσεων οι οποίες δεν θεωρούνται σωστές και δεν θα πρέπει να καταστέλλονται βία όπως έκαναν τώρα οι ε, κινέζικες αρχές. Τώρα διώχονται και εκτελούνται Ουιγούροι στη συνέχεια διαδηλώσεων μέσω της τυφλής χρήσης βίας από τον κρατικό μηχανισμό καταστολής. Θαυμάζουμε τον κινέζικο πολιτισμό Θαυμάζουμε την ικανότητά του στην επιχειρηματική, αλλά θα πρέπει να σηκώσουμε τη φωνή μας και να ακουστούμε καταδικάζοντας τις παραβιάσεις και τις εκτελέσεις. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις κινέζικες αρχές να τερματίσουν έστω και προσωρινά τις θανατικές εκτελέσεις και να ακολουθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενιαία πολιτική απέναντι σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Λόχ Μπίχλερ. Ευχαριστώ τις τελευταίες, ε, τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης για πολλούς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ε, τέτοιες ε, εξελίξεις θετικές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ποια θρησκευτική ή εθνοτική ομάδα προέρχονται. Αντιθέτως, οι διώξεις ουηγόρων και Θηβετιανών έχουν αυξηθεί σε ό,τι αφορά τη θανατική καταδίκη. Είναι θετικό το γεγονός ότι το Ανώτατο Κινέζικο Δικαστήριο από το 2007 ελέγχει πλέον ε, τις αποφάσεις αυτές για θανατικές καταδίκες και πλέον έχουν αναρρεθεί και κάποιες τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο, είναι πρωταθλήτρια η Κίνα στις εκτελέσεις. Το 2008 τουλάχιστον 1718 άτομα εκτελέστηκαν. Και με αυτό τον ε, ελάχιστο αριθμό, αν θέλετε, η Κίνα ευθύνεται για το 70% των εθνατικών ποινών σε όλον τον κόσμο. Οι Κινέζοι λοιπόν μπορούν πλέον να καταδικαστούν σε θανατική ποινή για περισσότερα από 68 εγκλήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό το ψήφισμα αυτό προκειμένου να υπάρξει ένα άμεσο μορατόριο σε ό,τι αφορά τις εκτελέσεις αυτές. μιλητές για πολιτικές ομάδες. Κύριος... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρότασή μου για την πρόταση ψηφίσματος ανήκει σε μια ιδέα ανθρώπου ο οποίος ε, ανήκει στις ιδέες ενός ανθρώπου που ανήκει σε μια τέτοια μειονότητα κέρδισε όμως το βραβείο Νόμπελ και βρίσκεται στην κορυφή μιας μεγάλης χώρας δύναμης, τον Ομπάμα. Αυτού οι αρχές είναι και δικές μου αρχές, αλλά δεν θα πρέπει να ξανακάνουμε τα λάθη της αριστεράς που θέλουν μόνο τα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά στο χαρτί. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και στην Κίνα όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλά πριν καταθέσουμε ένα τόσο σκληρό ψήφισμα, να έχουμε μια στρατηγική, ένα συντονισμό όλων των πολιτικών δυνάμεων και του συνόλου του Κοινοβουλίου για να μην επιμολύνουμε τις διαπραγματεύσεις με την Κινέζικη Δημοκρατία. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των μειονοτήτων και της θανατικής ποινής στην Κίνα χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το τι θέλει η κινέζικη κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό πράττει σωστά ο Ομπάμα, χωρίς να υποχωρήσει από τις αρχές του, διατηρεί σχέσεις με τις κινητικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει πρέπει να το παραδεχθούμε, να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον δυτικό κόσμο. Γιατί να, να καταθέσουμε ένα ψήφισμα λίγες ε, μέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής χωρίς σωστό συντονισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με την κυβέρνηση του Πεκίνου και πρέπει να μην βλάψουμε τις σχέσεις αυτές νέου τύπου με την κινέζικη κυβέρνηση. Συμμερίζομαι λοιπόν τις αρχές του ψηφίσματος, παρόλα αυτά θα τηρήσω θέση αποχής, γιατί νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό δεν θα βοηθήσει τη νέα σχέση που θέλουμε με την κινέζικη κυβέρνηση. Παρακαλώ την επόμενη φορά αν έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας να το σεβαστείτε. Σοσιαλιστές Γκόμες η Κίνα εξακολουθεί να καταπιέζει όλους αυτούς που διεκδικούν Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο κύριος Πόσελ θέλει το λόγο για διαδικαστικό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μας, η ομάδα μας είχε μετά από συζήτηση στην ε, συνέλευση των Προέδρων είχε ζητήσει αυτό το σημείο να έρθει στην μέση Ιδέα. Θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε θέλουμε να το ψηφίσουμε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν τώρα δεν ήταν η άποψη τη ομάδα μα, ήταν μια προσωπική άποψη του ομιλούντο. Το καταλαβαίνω κύριε Πόσελτ. Αλλά έχουμε ένα χρονικό διάστημα και η κάθε πολιτική ομάδα έχει ένα λεπτό για να παρουσιάσει την άποψή της. Εξακολουθεί η Κίνα να καταπιέζει και να καταστέλει όλους αυτούς που διεκδικούν κοινωνικά, πολιτικά, εργασιακά δικαιωμάτα, ακόμα και τα πιο βασικά. Η διάκριση αυτή ασκείται κυρίως κατά θρησκευτικών ομάδων και εθνοτικών μειοντήτων. Ο Χούτζα, βραβευμένος με το βραβείο Σάχαροφ, είναι ένας από τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται σε δίωξη μετά από την ε, τελευταία επίσκεψη του Ομπάμα στο Πεκίνο. Υπάρχει λοιπόν όλο και μεγαλύτερη καταστολή, όλο και μεγαλύτερη δίωξη των ε, ακτιβιστών. Όλα αυτά είναι τελείως σε αντίφαση με τις υποχρεώσεις της Δελακής Δημοκρατίας της Κίνας ως μέρους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ατόμων οι οποίοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Κίνα και έξω από την Κίνα. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι Κινέζοι είναι διαφορετικοί από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανμπάλεν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ως φιλελεύθεροι είμαστε κατά της αντικής καταδίκης, της αντικής ποινής γενικά. Αλλά εδώ στην Κίνα χρησιμοποιείται για την καταποίηση μειονότητας, μειονοτήτων όπως οι Ιγούροι οι Θεβετιανοί και έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δημοκρατία η Κίνα και δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει σκληρή πολιτική κατά της Τάιβαν. Θα πρέπει να ασκηθεί λοιπόν πίεση κατά της Κίνας. Είναι δύσκολο αυτό, το ξέρω, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις αρχές μας. Γι' αυτό λοιπόν και υποστηρίζουμε το ψήφισμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χουατάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό είναι μια σημαντική συζήτηση γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Και ένα τμήμα αυτής της συζήτησης θα πρέπει να είναι συζήτηση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε την υποχρέωση να υποστηρίξουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Τσιπάνκο να είναι σαφέ και να μπορέσουμε να τονίσουμε όλα αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια τη διάσκεψη κορυφή. Γι' αυτό δεν συμφωνώ με τον προηγούμενο συνάδελφο, ο οποίο ούτω και αλλιώ δεν με ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι, κατά, είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση στην Κίνα. Η Κίνα θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονό ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη παρά μόνο με μια διαφάνεια και με ένα σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και της ε, ελευθερίας της γνώμης. Μου φαίνεται πολύ παράξενο το ότι η Κίνα θέλει να αποκλίνει από αυτό το λόγο που είναι ο δρόμος που έχουν ακολουθήσει όλες οι δημοκρατικές χώρες του κόσμου. Μόνο με το σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η χώρα παγκόσμια τα ανθρώπινα δικαιώματα και οικουμενικά. Δεν μπορεί η Κίνα να είναι μία εξαίρεση. Και συμφωνώ με όλου αυτού που τόνισαν κάτι τέτοιο και πρέπει να αντιμετωπίσουν την Κίνα όπω και τι άλλε χώρε. Για τη συντηρητική ομάδα και τους ρεφορμιστές ο κ. Στάνοκ. εγώ πάντα άσκησα κριτική στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας Έχω διαμαρτυρηθεί επίσης και για τις διώξεις που υφίσταται η Ταϊβάν και την εκδίωξη της χώρας αυτής από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Έχω καταδικάσει επίσης και τις διώξεις της ειρηνικής τιβετιανής κουλτούρας, του Φαλουνγκόγκ, των χριστιανικών μειονοτήτων, των μέσων ενημέρωσης, του διαδικτύου και της Google. Καταδικάζω επίσης και τη διευρυμένη χρήση ε, της θανατικής ποινής όπως για την ε, για τη μαστροφία και τα οικονομικά εγκλήματα. Αν και για λόγους συζήτησης θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι, δικαιολογείται η χρήση της θανατικής ποινής, ορισμένα φρικτά εγκλήματα, δολοφονικά κτλ. Παρ' όλα αυτά, η λαϊκή δημοκρατία έχει εκφράσει την επιθυμία της να έχει πιο αρμονικές σχέσεις με τις εθνοτικές μειονότητες και ιδιαίτερα τους Ουιγούρους και άλλες μουσουλμανικές μειονότητες. Ζητώ επίσης να υπάρξουν και δίκες, δίκες για αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται. Κατσμαρεκ. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα του ΕΛΚΑ υποστηρίζει το σχέδιο ψηφίσματος. Ακούσαμε τις προτάσεις ε, ε, από πολλούς συναδέλφους ότι θα πρέπει σήμερα να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά μόνο για τη θανατική καταδίκη στην Κίνα. Έχουμε όμως την περχόμενη διάσκεψη κορυφής. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην δώσουμε στον πειρασμό και να εφαρμόσουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά κρατώντας και πάλι σιωπή μόνο και μόνο επειδή έχουμε έναν εταίρο που είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνουμε θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άσχετα αν έχουμε να κάνουμε με μια υπερδύναμη ή με μια μικρή χώρα όπω το Λάο ή το Βιετνάμ. Μπορεί να είναι μεγάλη χώρα, αλλά εκεί είναι ε, που γίνονται οι περισσότερες θανατικές εκτελέσεις. Δεν ε, κρατάει ούτε τα ελάχιστα προσχήματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδικασία δίκη δίκη αν ε, δεν ε, έχουμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια και να καταδικάσουμε τον κομμουνισμό, αν δεν είχαμε αυτό το θάρρος στην Ευρώπη, θα είχαμε τελείω διαφορετική μορφή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Παλέτσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι στον 21ο αιώνα θα καταργηθούν οι θανατικές ποινές και θα μείνουν μόνο στα μουσεία ε, οι συσκευές που εφαρμόζονται, που χρησιμοποιούνται για την ε, θανατική εκτέλεση των κατηγορουμένων. Η Κίνα δεν είναι μόνο η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή και το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και χώρα που έχει τις περισσότερες θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις. Βέβαια, πολλοί θα πούνε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Αν όμως μιλούμε για στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, που είναι σημαντική και για τις δύο πλευρέ, θα πρέπει να ζητήσουμε από το Πεκίνο να αλλάξει την πολιτική του ω προς τη θανατική ποινή, αλλά και ω προς το διάλογο με τις εθνοτικές μειονότητε. και να προκρίνει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Κυρία Λεχτενμπεργκεν, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί ένα διαρκές θέμα σύγκρουση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λαϊκής Δημοκρατία τη Κίνα. Η κατάσταση των ε, μειονοτήτων χειροτερεύει ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ω εκ τούτου διαπιστώνουμε ότι το Θιβέτ και οι Ουιγούροι τίθενται υπό περισσότερη πίεση τους τελευταίους μήνες. Άρα δεν καταλαβαίνω το γεγονός ότι θέλουμε να αφαιρέσουμε το σημείο 9 από το ψήφισμα, γιατί για παράδειγμα μιλάμε για ειρηνικό διάλογο αντί για καταπίεση. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός ε, φορέας στην διεθνή σκηνή αλλά θα πρέπει να επιδείξει την απαραίτητο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό δεν αναφέρεται, δεν φτάνει ε, να αναφέρεται αυτό στο Σύνταγμα, θα πρέπει και συγκεκριμένα να εφαρμόζονται, να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Θηβετιανών, των Ιγούρων και των άλλων μειονοτήτων στην ε, Κίνα. Ευχαριστώ κύριε Λέχτενμπεργκερ. Ο κύριος Πόσελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Το έχω πει ήδη μία φορά. Στο κέντρο των ελεύθερων Ουιγούρων. Για τον ίδιο λόγο που και ο πρόεδρος έχει δραστηριοποιηθεί υπέρ των Τσέχων πριν από κάποια χρόνια, γιατί εκεί ήταν το κέντρο των ελεύθερων δικαιωμάτων, αν θέλετε. Και αυτή η πνευματική ελευθερία υπάρχει σήμερα ακόμα. Παράλληλα, ο Στράους, ο οποίος ε, πάντα υπεράσπιζε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, ε, υποστήριξε τις ε, ελεύθερες σχέσεις μας με την Κίνα. Δεν αποκλείει το εν το άλλο όμως να έχουμε καλές επαφές με την Κίνα, αλλά και παράλληλα να έχουμε σαφή θέση σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά και λοιπά ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν αυτή την εβδομάδα έγιναν διάφορες επιχειρήσεις σκούπες στο Μόναχο όπου συνελήφθησαν Κινέζοι αξιωματόχοι που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παρακολουθούν και να τρομοκρατούν τους τους Ιγούρους αυτό καταδεικνύει τι μεθόδους χρησιμοποιεί η Κίνα. Αυτές τις μεθόδους δεν μπορούμε να τις ε, αποδεχτούμε γιατί ξεκινάνε από τέτοιες τρομοκρατικές ουσιαστικές οργανώσεις, ε, δράσεις στο Μόναχο και κορυφώνονται σε θανατικέ καταδίκες στην Κίνα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πίτσι. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει για να σώσει ανθρώπους από τη θανατική ποινή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές και όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα μορατόριο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, για την μη εκτέλεσμα της θανατικής ποινής. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι πρόσχημα για να κατηγορήσουμε την Κίνα για να θέσουμε την ε, ακεραιότητα της Κίνας σε αμφισβήτηση ή να κάνουμε μια καρικατούρα της Κίνας. Δεν βοηθάμε τους ανθρώπους στην Κίνα που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και την κοινωνική αρμονία όταν εμείς δρούμε με αυτόν τον τρόπο. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους προσπαθήσουμε να τους ε, επιμορφώσουμε με τις λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες. Δεν μπορούμε τώρα με ένα θέμα κατεπήγοντος, με ένα ψήφισμα κατεπήγοντος, να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το μνημόνιο για την ελευθερία του λαού του Θιβίτ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ελευθερίες των λαών, ούτε αποτελεί μια αποδεκτή θέση. Ελπίζω ότι στο μέλλον ότι θα είναι η τελευταία φορά που πριν από μια διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα γίνεται μια τέτοια συζήτηση κατεπήγων και δεν γίνεται μια ευρεία συζήτηση η οποία θα αντιμετωπίσει όλο το φάσμα των ζητημάτων που έχουμε να κάνουμε με την Κίνα. Ευχαριστώ. Ήταν μακρηγόρησε τελικά και άλλα πολλά αυτά. Ο κύριο Σούλτ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριο Μπούτι Κόφερα. Η ειδική μου πολιτική ομάδα είχε ζητήσει εμείς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επαπειλούμενης θανατικής ποινή κατά των Ουιγούρων στην Κίνα και το γεγονός ότι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο αυτοί που έλαβαν μέρος σε ε, διαδηλώσεις ειρηνικές κατά των εκλογών, του αποτελέσματος των εκλογών, των φαλκιδευμένων εκλογών στο Θιβέτ. Επομένως το κατεπήγον αφορούσε την επαπειλούμενη ποινή θανάτωσης ορισμένων ανθρώπων. Το ότι οι Κινέζοι έχουν ρεκόρ θανατικών εκτελέσεων και ότι είναι ένα κράτος το οποίο καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Αλλά εμεί ζητήσαμε στην συζήτηση των αρχηγών των πολιτικών ομάδων να συζητήσουμε το κατεπήγον, δηλαδή τις θανατικές ποινές και το συνολικό θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε πολιτιστικό, σε επίπεδο εξοπλισμών να τα αντιμετωπίσουμε σε μια χωριστή συζήτηση για τη διάσκεψη κορφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και όχι μέσα σε ένα ψήφισμα κατεπήγοντος. Γι' αυτό ε, θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το κατεπήγον εμείς πρέπει να ψηφίσουμε το θέμα του κατεπήγοντος και όχι να μιλήσουμε για όλο αυτό το, το συνονθήλευμα από απόψη σε σχέση με την Κίνα. Διαδικασία catch the eye. Catch the eye για δύο λεπτά. Θα δώσω το λόγο σε ένα ομιλητή από κάθε ομάδα. Οι σοσιαλιστές μόλις έλαβαν το λόγο. Από το και έχει το λόγο ο κύριος Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και είναι σημαντικό το, οποίο, το γεγονός ότι αυτό το θέμα ήρθε στα κατεπήγοντα και μάλιστα με πρωτοβουλία τσέχων ε, Ούγγρων ε, πολιτών. Αυτό καταδεικνύει ότι υποστηρίζουμε και το συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία. Μου προκαλεί κάπω έκπληξη το γεγονό ότι οι σοσιαλιστέ τώρα κάνουν ένα βήμα προ τα πίσω, επαναχωρούν σε σχέση με την πρόταση αυτή ψηφίσματο. Με λυπεί ιδιαίτερα αυτό. Με λυπεί και γιατί το κείμενο αυτό επί του οποίου συμφωνήσαμε προχτές δεν έχει πλέον καμία αναφορά σε κομμουνιστικά καθεστώτα και καμία αναφορά σε λεπτομέρειες και σε στοιχεία αναφορικά με την προστασία των μειονοτήτων. Θεωρώ ότι είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με αυτά που έχουν αφήσει πίσω τους ο κομμουνισμός και μάλιστα με ανοιχτό τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Μάιστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι σαφές ότι είμαστε κατά της θανατικής ποινής όπου και να πρόκειται σε όλο τον πλανήτη μας. Και είμαστε εναντίον τη καταπίεση οποιασδήποτε μειονότητας και όχι μονάχα των Ουιγούρων. Αλλά και τα δύο συμβαίνουν στην Κίνα. Πολλά έχουν γίνει με ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων πέρσι. Επειδή είναι γνωστό για τους Κινέζους ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση τη Κίνα. Αυτό ελπίζαμε θα οδηγήσει σε λιγότερα, λιγότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ είναι το αντίθετο. Έχουμε όλο και περισσότερε εκτελέσεις και εμείς έχουμε την περίπτωση των Ουιγόρων. Πολλοί από αυτούς έχουν εκτελεστεί και επίσης ίδιες απειλέ ασκούνται κατά των Θηβετιανών. Η Κίνα μπορεί να είναι ένα σημαντικό ε, εμπορικό εταίρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο και αν είμαστε αμήχανοι ενώπιον λοιπόν σε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα μέσα στην ημερήσια διάταξη τη ε, διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα και γι' αυτό είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει να υπάρξει εφαρμογή του μορατόριου που είχε ζητηθεί το 2007 για τη θανατική ποινή και να μην εκτελεστούν άλλε θανατικέ ποινέ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ευχαριστώ. Ως Πολωνός αισθάνομαι πάντα να σκυρτάω, να χτυποκαρδώ κάθε φορά όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί οι Πολωνοί το 1989 είχαν τις πρώτες εκλογές από τις οποίες προέκυψε ε, μη κομμουνιστής πρωθυπουργός. Ενώ εκείνη την ίδια χρονιά η Κίνα με τα τεθωρακισμένα ε, καταπίεσε και σκότωσε πολλούς φοιτητές που διαδηλώναν στην πλατεία Μεν. Μετά από χρόνια η Ευρώπη κατάφερε να νικήσει τον Σοβιετικό κομμουνισμό. Δυστυχώς δεν κατάφερε εκείνα να καταπολεμήσει τον κομμουνισμό. Και είχε συστηθεί από πολλές χώρες ότι θα μποϊκοτάρουν την ε, εναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων. Δυστυχώς ε, ε, πριτάνευσαν κάποια εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα και κανένας δεν τόλμησε να μποϊκοτάρει εκείνη την τελετή των, των, των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Δεν έχουμε μόνο τη θανατική ποινή, αλλά έχουμε βασανιστήρια, φυλακίσεις, ε, φήμωση της ελευθερίας έκφρασης, ε, της ελευθεροτυπίας. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό το ψήφισμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πρετανεύσουν οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αξίες της ανθρώπινης ελευθερίας έναντι των εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων. Το λόγο έχει τώρα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Δεχούχτ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να εξηγήσω πώ έχουν τα πράγματα μεταξύ των σχέσεων, σε σχέση μεταξύ Κίνα και Ευρώπη. Η πολιτική μα είναι μια πολιτική επικοδομητική εμπλοκή. Είμαστε δύο μείζονες εταίροι στην παγκόσμια σκηνή, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Στις 30 Νοεμβρίου στο Ναντζίνγκ θα γίνει η συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας. Θα συζητήσουμε τα θέματα της συνάντησης της Κοπενχάγης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική κρίση και όλα τα διεθνή θέματα. Η στρατηγική αυτή σχέση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο τα πάντα. Είναι σαφές ότι η Κίνα και η Ευρώπη μπορεί να έχουν διαφορές σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Η δύναμη όμως της σχέσης μας μας δίνει τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θανατική ποινή και τα δικαιώματα των μειονοτήτων τίθενται συστηματικά κατά τη διάρκεια των τακτικών επαφών που έχουμε και στα πλαίσια του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις κινέζικες αρχές. Αυτό έγινε και κατά στις 20 Νοεμβρίου στο Πεκίνο. Είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά η, η αντίθετη άποψη, ε, άποψή μας μάλλον, η αντίθετη με τη, τη θανατική ποινή ε, τίθεται συνεχώς, όπως επίσης και το θέμα του σεβασμού των μειωνοτικών ε, μειονοτικών δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να θέτουμε τα θέματα αυτά και σε διαφορετικά φόρα, στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Η συνάδελφος Φερέρα Βάλνερ είχε το Μάρτιο που πέρασε μια πολύ σημαντική συζήτηση με τους Κινέζους, υπογράμμισε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογραμμίσω εδώ, να θυμίσω κάποια από τα στοιχεία της πολιτικής μας. Πάντα υποστηρίξαμε τον διάλογο ανάμεσα στις, κοινοτικές, στις κινέζικες συγγνώμη, αρχές και τους εκπροσώπους του Δαλάη Λάμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι καθολικά θεμελιώδη και στο Θιβέτ και είναι βασική ανησυχία της διεθνούς κοινότητας. Η κατάσταση στο Θιβέτ συστηματικά αντιμετωπίζεται με αυτή την αντίληψη. Έχουμε στείλει το μήνυμα αυτό στους Κινέζους ομολόγους μας και έχουμε ακούσει στις απαντήσεις τους προσεκτικά. Η Επίτροπος Άστον τον Ιούλιο εξέφρασε τις ανησυχίες της για την κατάσταση στο Σινγιάνγκ, η οποία προκάλεσε πολλούς θανάτους και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση, ε, για την συμφιλίωση μάλλον των εθνοτήτων στην περιοχή αυτή. Επιβεβαιώνουμε επίσης την καθολική μας αντίθεση στη χρήση της θανατικής ποινής κάτω από οιασδήποτε συνθήκες και τη σημασία που δίνουμε εμείς στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τις ανησυχίες της επανειλημμένα προς τις κινέζικες αρχές και το έκανε αυτό και στις δύο δηλώσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 29 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου. Όπως πάντα γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι δηλώσεις αυτές καλούν την Κίνα να μετατρέψει όλες τις θανατικές ποινές που έχουν σχέση με τις με τις ε, ταραχές στο Σινκιάν και στο Θιβέτ και να μην χρησιμοποιήσει τη θανατική ποινή σε ε, αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια πιο ε, δεκτική και ανοιχτή Κίνα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον τομέα της υπεπίδησης των διεθνών προκλήσεων. Νομίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες, ελπίζαμε μάλλον, θα ήταν η αρχή μιας μεγαλύτερης ευελιξίας στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων και κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της στρατηγικής μας στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι αναπόσπαστο τμήμα του συνεχούς διαλόγου. Η συνάντηση κορυφής του Πεκίνου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προχωρήσουμε στην εξέλιξη περαιτέρω των σχέσεών μας. Ευχαριστώ Επίτροπε. Αυτό είναι το τέλος της συζήτησης για την Κίνα και τώρα θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Έχουμε τρεις προτάσεις για την Ικαράγουα. Έχει ζητήσει το λόγο η Ντεκεζέρ η ομάδα μας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ψηφοφορία για τους λόγους που ανέφερε